Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά την πολύ εντατική πρωινή συνεδρίαση και τη χθεσινή, επίση εντατική, περνάμε στο τρίτο κομμάτι τη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας που προβλέπει την παρουσίαση κάποιων καταξουσιοδότηση πράξεων από τον Διευθυντή Γιάνς Σχάπς. Καλωσορίζω θερμότατα τον Διευθυντή και τους εκπροσώπους ε, της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη. Η κατεξοδότηση πράξεις αφορούν την κοινή οργάνωση αγοράς και τις σχετικές ε, πράξεις που πρέπει να υιοθετηθούν μέχρι τον Νοέμβριο του 2015. Η δέσμη προβλέπει τέσσερι καταξιδότηση ε, κανονισμού, τον κανονισμό για τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση ιδιωτική αποθεματοποίηση, τη κοινοποίηση των κρατών μελών και τη διαδικασία μετάδοση πληροφοριών για τι άμεσε ενισχύσει και πτυχέ που αφορούν τι γεωργικέ αγορέ, Επίσης, εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων των οργανισμών, οργανώσεων παραγωγών και διακρατικούς και διακλαδικούς ε, και θέματα διακλαδικών και διακρατικών ε, οργανισμών και άδειες ε, εισαγωγών-εξαγωγών. Για όλα αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει κατεξοδότηση πράξης στα πλαίσια της προσπάθειας απλούστευσης της διαδικασίας. Έχετε λάβει σχετικό υλικό και τεκμηρίωση. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη, τον Διευθυντή, τον κύριο Γιένς Σχάπς, που θα μας παρουσιάσει τις τέσσερις αυτές καταξιοδότηση πράξεις. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ σήμερα εδώ μαζί σας, έτσι ώστε να σας δώσω τα πρώτα αποτελέσματα της ε, εργασίας που έχουμε ολοκληρώσει τους τελευταίους ε, μήνες σε συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα πλαίσια των ομάδων εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τον κανονισμό ε, για το, μάλλον την ευθυγράμμιση των ε, κανονισμών για την κοινή οργάνωση αγοράς ε, με την συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει να σας πω ότι και ο Γενικός μου Διευθυντής πολλές φορές ήταν στην Επιτροπή σας έτσι ώστε να εκφράσει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να οργανώσει την εργασία της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 200 κανονισμούς εκτελεστικούς που πρέπει πλέον να γίνουν κάτι πιο ολοκληρωμένο και ενοποιημένο ε, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει πλέον η συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά τις κατεξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Ε, έτσι θέλουμε επίσης να πλουστεύσουμε τους υφιστάμενους ε, ε, κανονισμούς έτσι ώστε να μειώσουμε τον, το ποσοστό λάθους των αγροτικών δαπανών, να αυξήσουμε την συνεκτικότητα της πολιτικής μας, να, να γνωστοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και τέλος να οδηγηθούμε σε αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα και αυτό στο σύνολο τη διαχείριση της γεωργικής αγοράς. Μέχρι τώρα έχουμε ε, κάνει κάποιες ε, τροποποιήσεις, κυρίως όσον αφορά ε, το, την ε, καταπολέμηση της λευκής μήγας του ελαιολάδου, καθώς επίσης και το, τις αδειοδοτήσεις φύτευσης στο εμπελοϊνικό τομέα, που έχει και αυτό ολοκληρωθεί. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν το, πρώτη, το πρώτο τμήμα της τη δέσμης απλούστευσης και γι' αυτό έχουμε υποβάλει ε, και τις ε, ε, προτεραιότητες που ανέφερε ο πρόεδρος προηγουμένως, ιδιωτική αποθήκευση, εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων των οργανώσεων, άδειε εξαγωγών εισαγωγών, καθώς επίσης και κοινοποιήσεις στοιχείων από τα κράτη-μέλη υπό το σύστημα ΙΣΑΜ. Επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα ε, είναι μια άλλη δέσμη που θέλουμε να σας παρουσιάσουμε λοιπόν, αλλά επισύνοντας την προσοχή σας ότι εδώ έχουμε μόνο το πρώτο τμήμα ε, και θα ακολουθήσουν και άλλα. Στους επόμενους μήνες ε, θα ακολουθήσουν και άλλα στοιχεία και τους πρώτους μήνες βέβαια του 2016 για λαχανικά την, ε, τις ετικέτες, τη σήμανση, ε, ε, τη διαχείριση τη, των οργανώσεων ε, αγοράς, τη διαχείριση κάποιων κατεξουσιοδότηση πράξεων όσον αφορά την ρύθμιση, τους ε, κάποιους κανόνες ρύθμισης της αγοράς και ε, της, εμπορίας. Αυτό θα γίνει μέχρι την αρχή του 2016. Ας επανέλθουμε όμως στις Βουλίες που θέλουμε να σας παρουσιάσουμε, κυρίως έτσι ώστε να σας ε, ε, επιστήσουμε την προσοχή σε κάποια σημεία τα οποία, ε, με τα οποία ασχολείστε ήδη και εσείς για να σας δώσουμε μία σύνοψη λοιπόν από τεχνική άποψη τι έχουμε κάνει και για να μπορέσουμε να έχουμε και από τη δικιά σας πλευρά κάποια σχόλια και κάποιες δικές σας σκέψεις όσον αφορά ε, τις προτεραιότητες αυτές. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα στην ενίσχυση για τη δημόσια παρέμβαση και την ιδιωτική αποθήκευση. Έχουμε αυτή τη στιγμή έξι ε, κανονισμούς εφαρμοστικούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε με τις υφιστάμενες τεχνικές παραμέτρους ε, με κάποια εξαίρεση όσον αφορά τα πρωτεϊνούχα, όσον αφορά ε, τα, τα δημητριακά. Ε, επίσης θα δούμε το θέμα της ζάχαρης και πιο εξειδικευμένα τις κάποιες ειδικές ποσότητες οι οποίες έχουν αντιμετωπιστεί με διαφορετικές δυνατότητες αποθήκευσης με την δική σας ε, συμμετοχή έχουμε βρει ε, κάποιες λύσεις όσον αφορά την ε, αποθήκευση και έχουμε προχωρήσει αρκετά, έχουμε συνεργαστεί με όλα τα κράτη-μέλη και όσον αφορά την επιλεξιμότητα των φορέων, των operators, ε, θα πρέπει να ε, έχουμε συμφωνήσει ποιες είναι οι ποσότητες οι οποίες θα μπαίνουν, θα στέλνονται στην ε, παρέμβαση. Αυτό είναι λίγο, είναι λίγο διαφορετικό σύστημα από αυτό που είχαμε στο παρελθόν. Όσον αφορά τώρα την εξωτερική ανάθεση του outsourcing, καθώς επίσης και την Διεθνική Συμφωνία, η εξωτερική ανάθεση ε, κυρίως ε, όσον αφορά η, ε, και τις του εκδοσιακούς οργανισμούς έχουμε κάποιες νέες αρχές όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων, την αρχαιοθέτηση καθώς και εδώ έχουμε μια επιπλέον ευελιξία, οι εξειδικευμένους κανόνες όσον αφορά την αναγνώριση των ε, των οργανώσεων των παραγωγών αλλά και των διακλαδικών ε, οργανώσεων σε διεθνές επίπεδο όπου θέλουμε να καταστεί σαφές ότι τα κράτη-μέλη ε, μπορούν να αναλάβουν την πρωτοβουλία αναγνώρισης των οργανισμών αυτών. Τέλος, με αυτήν την διαδικασία έχουμε βάλει τρεις ε, τομεακούς ε, εκτελεστικούς ε, κανονισμούς για το καπνό uh, um, και για δύο άλλα είδη. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα των αδειών για τις εισαγωγές και εξαγωγές των γεωργικών προϊόντων ε, θα θέλαμε ε, ε, να υπάρχει ενιαίο νομικό πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει τους τρεις συν έξι εφιστάμενους κανονισμούς και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι για όλα τα προϊόντα ε, τα, για τα οποία υπάρχουν ποσοστώσεις ε, καθώς επίσης ε, και άδειες για προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγών αυτά διατηρούνται. Ο αριθμός των προϊόντων τα οποία υφίστανται αδειοδότηση, να πούμε ότι αυτές οι άδειες λειτουργούν μονάχα σαν εργαλείο επιτήρησης, διότι εντωμεταξύ ε, έχουμε ε, βρει πολύ πιο αποτελεσματικούς τρόπους έτσι ώστε να ε, μετρούμε, να υπολογίζουμε τις εισαγόμενες ποσότητες κυρίως μέσω του συστήματος επιτήρησης της ταξίδ και είναι ένα σύστημα το οποίο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ε, και έχει γίνει πλέον ένα πολύ ισχυρό αλλά και αξιόπιστο εργαλείο από τη δική μας σκοπιά τουλάχιστον. Ε, οι άδειε και αυτό θα είναι ο αντίκτυπος ε, θα περιοριστούν μονάχα σε εισαγωγές με καθεστώς προτιμησιακό και θα περιοριστούν σε ορισμένα κρίσιμα ε, ε, προϊόντα όπως είναι ας πούμε η ε, ζάχαρη και κάποια άλλα όσον αφορά uh, the uh, false classification in the common όλα αυτά βέβαια τα βλέπουμε και υπό το καθεστώς της, ε, της ονοματολογίας και σε στενή συνεργασία με την Όλαφ διότι το σύστημα ε, αδειοδότησης ενδεχομένως δεν είναι ο καλύτερος τρόπος έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η ε, απάτη. Αυτό που θέλουμε ε, είναι να δούμε τι δυνατότητες έχουμε στα σιτηρά τουλάχιστον έτσι ώστε να καταφέρουμε να επιτύχουμε ένα σύστημα επιτήρησης που να είναι πιο πιο ισχυρό, βασιζόμενο πάντα στο σύστημα ταξίδ ε, και ε, το reporting να γίνεται κάθε εβδομάδα και όχι κάθε μήνα. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στο τελευταίο εργαλείο, το οποίο είναι η μετάδοση ε, των πληροφοριών ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών και στοιχείων από τα κράτη-μέλη. Εδώ το κυριότερο θέμα ε, είναι ότι οριστικά θα διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, δεν θα χρειάζεται ε, να επιστρέφουν τις μηδενικές ή κενές κοινοποιήσεις ε, και με τον τρόπο αυτό θα μειώσουμε αισθητά τον αριθμό και τον όγκο των πληροφοριών ε, που στέλνουν τα κράτη-μέλη. Ε, αυτό μας το επιτρέπει το σύστημα διαχείρισης και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας. Τέλος, από τη δική μας πλευρά είμαστε ε, πολύ ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί μέχρι τώρα. Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων ε, αποτέλεσε ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Νομίζω λοιπόν ότι ε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε ε, τη συνεργασία επί των συγκεκριμένων νομικών κειμένων συγγνώμη, ε, τα οποία θα είναι οπωσδήποτε πολύ πιο συγκεκριμένα από ό,τι τα τεχνικά δελτία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό ήθελα να πω και σίγουρα μπορείτε να μας υποβάλλετε οποιαδήποτε ερώτηση και είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Πρώτος θα λάβει το λόγο ο βασικός μας συζητητής για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωρικής πολιτικής για την περίοδο 2014-2020 και ιδιαίτερα για το θέμα της κοινή οργάνωσης αγορών, ο κύριος Νταντά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Νταντά. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την παρουσίασή της. πάμε. Πραγματικά και για άλλη μια φορά εκφράζω ότι μου γιατί δεν υπάρχουν επαφές μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών πριν να δημοσιευθούν τα κείμενα για τις κατεξουσιαδότηση πράξης. Η δυσκολία που επικρατεί στην αγορά είναι εμφανής. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο είναι τελικά η αποθήκευση, η αποθεματικοποίηση και αυτό που βλέπουμε είναι αν ε, μπορεί κανείς να μιλήσει για περίληψη των διαφόρων κειμένων θα έλεγα ότι απλοποίηση δεν θα πρέπει να σημαίνει απαραίτητα και θυσίες. Διότι κάθε φορά που μιλάμε για απλοποίηση θα πρέπει να ζητάμε την αποτελεσματικότητα στην πράξη και όχι μόνο την εξάλληψη της γραφειοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο και έχοντας αυτό κατά νου, πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα κοιτάμε όλες αυτές τις απόπειρες απλοποίησης, τουλάχιστον από εδώ και πέρα. Τώρα, η μεταφορά δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και αυτή η διαδικασία απλοποίησης. Βεβαίω αυτό που δημιουργήσαμε στην αγορά του γάλατος με το παρατηρητήριο ήταν να υπάρχει αξιόπιστη και ταχεία μεταφορά δεδομένων. Διότι περάσαμε από την περίοδο που δεν έπρεπε να μας απασχολήσει η αγορά, διαπιστώσαμε ότι εάν εμείς δεν ασχοληθούμε με την αγορά, δυστυχώς εμείς, εμείς ενώ οι Ευρωπαίοι, θα είμαστε αυτοί που θα πέσουμε στην παγίδα. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε οι νέες τεχνολογίες να μην είναι χρονοβόρες, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς επιτόπου και έτσι όταν έρχεται η Επιτροπή και μας προτείνει μια κατάσταση για την αγορά να μπορεί να μας μιλήσει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κοντά σε μας και όχι πριν από χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν βελτίωση της κατάστασης και σήμερα χάρη στο παρατηρητήριο για το γάλα διαθέτουμε πληροφορίες πάρα πολύ ενημερωμένες για το για την αγορά αυτή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα και περιμένω να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση. Έχω μια σύσταση, μια συμβουλή προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν λαμβάνει πληροφορίες από τα κράτη-μέλη και δυστυχώς ε, το παράδειγμα της πατρίδας μου είναι μάλλον αρνητικό σε ό,τι αφορά την κοινοποίηση δεδομένων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα θέμα δηλαδή που είναι συναφέ με το φλέγον ε, ζήτημα που συζητούμε σήμερα, η τιμή του γάλακτος. Ε, η τιμή που ενήγγειλε η κυβέρνηση υπερβαίνει κατά τα 22 λεπτά το, το λίτρο. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει 0,10 ε, για την ε, Ρουμανία. Δεν θα πρέπει να στηρίζετε, να στηρίζετε μόνο σε κυβερνητικές ε, πηγές και πληροφορίες άσχετα από ποια παράταξη προέρχονται οι κυβερνήσεις. Θα πρέπει να έχετε άμεσες επαφές με, τους, με τις οργανώσεις παραγωγών, γιατί αυτοί έχουν τα πραγματικά και ακριβή στοιχεία. Μην στηρίζετε μόνο στις κυβερνητικές πληροφορίες. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κούσμιουκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Διευθυντή για την παρουσίαση και την ενημέρωση. Ως εκπρόσωπος όμως μια μεγάλης σχετικά νέας χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Πολωνίας, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν αυτό το εθνικό κονδύλιο που αφορά τη στήριξη των παραγωγών ε, κρέατος που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είναι τόσο πενιχρή. Ούτε 29 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι για μας. Ούτε 7% δηλαδή του συνολικού κονδυλίου για τη στήριξη των κτηνοτρόφων. Και βλέποντας την κατάσταση στη χώρα, διαπιστώνω ότι η παραγωγή γάλακτος και κρέατος έχουν προβλήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά στην Πολωνία είχαμε και φοβερή ξηρασία. Κάτι που μας κατέστρεψε. Και είχαμε ραγδαία μείωση των συγκομιδών και στα φυτά και θα έχουμε πρόβλημα και στην ε, εκτροφή γιατί έχουν ξεραστεί οι βοσκότοποι και θα χρειαστούν μερικοί κτηνοτρόφοι να σφάξουν κοπάδια γιατί δεν μπορούν να τα θρέψουν. Οπότε η πενιχρή βοήθεια και στήριξη που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να καλύψει ε, τους Πολωνούς Γεωργούς. Μάλιστα και το Υπουργείο Γεωργίας Πολωνίας ε, πρόβλεψε στήριξη, αλλά και αυτή είναι συμβολική. Γιατί λοιπόν ε, ε αντιμετωπίζετε την Πολωνία τόσο δυσανάλογα σε σχέση με το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Πολωνοί Γεωργοί για κτηνοτρόφοι. Ευχαριστώ. Μάλιστα, άλλο κανεί. Δεν ζήτησε άλλο κανείς το λόγο. Α, ο κύριος Μπούντα πάλι. Μία ακόμη σκέψη, μία Συμβουλή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς ε, θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη. Πρόσφατα έχει μοιράσει 500 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία, αλλά δεν χρειάζεται μόνο να, να σκορπάτε κονδύλια. Θα πρέπει να εξακριβώνετε κατά πόσο αυτά τα χρήματα φτάνουν στους άμεσα ενδιαφερομένους, στους ε, γεωργούς. Τα 11,4 εκατομμύρια που εστάλησαν στη Ρουμανία, από τα 11,4, τα 3 ή 4 εκατομμύρια θα τα πάρουν εταιρείες που προωθούν ε, τα ρουμανικά προϊόντα, όχι η ίδια παραγωγή. Σας ενδιαφέρει ποιοι είναι οι πραγματικοί παραλήπτες αυτής της βοήθειας, γιατί καλό είναι να την επιταψιλεύετε, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε αν φτάνει στα σωστά χέρια. Ευχαριστώ. άλλο κανείς? Όχι. Οπότε να κάνω κι εγώ κάποια σύντομα σχόλια. Γενικώ. θεωρώ ότι ελάχιστη προσοχή δίνουμε στο θέμα της οργάνωσης αγοράς και αφιερώνουμε πενιχρά κονδύλια στην παρέμβαση. Κάτι που προκαλεί αστάθεια και ανησυχεί και προβληματίζει τα μάλα τους Γιώργους. Γι' αυτό και είχαμε, οι Γεωργοί είχαν πολύ ψηλές προσδοκίες γιατί η γεωρική παραγωγή έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες και πολύ μεγάλες διακοιμάνσεις. Και φυσικά οι διακοιμάνσεις στην παραγωγή προκαλούν αστάθεια και στην αγορά εξαιτία και της αστάθειας των τιμών. Η πείρα μας μας έχει δείξει ότι είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στις κατεξουσιοδότηση πράξεις γιατί συχνά μας ευνηδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις λύσεις που προτείνει στις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Γι' αυτό και είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί. Θα προτιμούσαμε να έχουμε πιο τεκμηρωμένη ενημέρωση και πιο έγκαιρη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις λύσεις που προτείνει στις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Και δεν θα πρέπει οι λύσεις αυτές να αποκλίνουν από την κατεύθυνση που δίνουν οι βασικές νομοθετικές πράξεις. Βέβαια ξέρουμε ότι η ζωή είναι περίπλοκη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να διασφαλίσει την επιρροή της, την επιρροή που είχε μέχρι τώρα όταν ο επιμερισμός των ρόλων μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων ήταν διαφορετικός και προσπαθεί και η Ευρωπαϊκή Επιρροή να κρατήσει την επιρροή της, αλλά και εμείς έχουμε ιδιαίτερες ευαισθησίες. Γι' αυτό και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις δικές μας, και τις δικές μας προτάσεις και συστάσεις. Αυτά κύριε Διευθυντά. Θα σας ξαναδώσω το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Σας ακούμε. Thank you. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω σε ορισμένες από τις ερωτήσεις, όχι σε όλες, γιατί δεν αφορούν όλες το ε, πλαίσιο της συζήτησης αλλά και των αρμοδιοτήτων μου. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την συνεργασία με τα κράτη-μέλη ε, καθώς επίσης να διευκολύνουμε και την μετάδοση των ε, στοιχείων και εδώ ο κύριος Νταντών βεβαίως έπιασε στόχο γιατί είδαμε προσπάθειες της Κομισιόν και στο παρελθόν έχουν ξεκινήσει κάποιες δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ικανότητα συλλογής στοιχείων, ανάλυσης της αγοράς με στοιχεία τα οποία ε, είναι πρόσφατα, μας φτάνουν γρήγορα, είναι αξιόπιστα ε, και επομένως μπορούμε να τα αναλύσουμε καλά. Το σύστημα ΕΣΑΜΑ είναι ένα σύστημα το οποίο ε, χρησιμοποιείται για αυτόν ακριβώς τον σκοπό και μάλιστα ε, πηγαίνει ακόμα πιο πέρα από το στενό πλαίσιο των κατεξουσιοδότηση πράξεων μπορούμε, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα στοιχεία τα οποία μας φτάνουν ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία μας ε, με ταχύτητα και ασφάλεια και αξιοπιστία βεβαίως, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Φυσικά το αποτέλεσμα εξαρτάται και από την ποιότητα των στοιχείων που μας θέλουν τα κράτη-μέλη, ε, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρά τα στοιχεία που μας φτάνουν από τα κράτη-μέλη. Είναι γεγονός ότι για κάποιες αγορές οι καθυστερήσεις που ε, σημειώνονται είναι μεγαλύτερες από ό,τι θα επιθυμούσαμε. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε και την ε, ε, ορθότητα των στοιχείων και την ταχύτητα. Όσον αφορά τώρα τις πληροφορίες που έχουμε Χρησιμοποιούμε και το σύστημα εποπτείας ε, και επιτήρησης ε, ταξίδ, το οποίο είναι όλο και πιο αξιόπιστο. Ε, εκεί καταλήγουμε λοιπόν μετά από οκταετή εμπειρία. Και για την ώρα αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι το σύστημα είναι πολλά υποσχόμενο, έχουμε στοιχεία τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στην πραγματικότητα, και ε, σίγουρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο και περισσότερο και ε, όλο και πιο αποτελεσματικά αυτά τα στοιχεία ε, για λόγους εμπορίου. Κύριε Πρόεδρε, και σε σχέση με αυτό που είπατε και εσείς μόλις τώρα, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εμπλέξουμε όλους τους φορείς όλους όσοι έχουν ενδιαφέρον για τον τομέα αυτό και βεβαίως για μία ακόμα φορά θα επαναλάβουμε ότι το Κοινοβούλιο είναι ευπρόσδεκτο στις ε, συζητήσεις μας και ότι επανειλημμένα και το τεχνικό μας προσωπικό έχει συζητήσει για τα θέματα αυτά ε, στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία γιατί έπεται ε, ε, αντιμετώπιση πολλών άλλων θεμάτων στο μέλλον και νομίζω ότι όλοι όσοι συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία ε, όλοι λοιπόν έχουν την άποψη ότι πρόκειται για μια διαδικασία ανοιχτή η οποία δίνει στον καθένα την δυνατότητα να εκφράσει τον προβληματισμό του και μάλιστα αυτό αποδεικνύεται και από την σημερινή μας παρουσία εδώ γιατί πραγματικά θέλουμε να συζητήσουμε σε βάθος όλα τα ε, ζητήματα και αυτό σημαίνει και αυτό αποδεικνύει μάλλον πόσο σοβαρά ε, λαμβάνουμε υπόψη το διάλογο αυτό. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες απορίες και ερωτήσεις, να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή, τον κύριο Σχάπς, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενημέρωση που μας έκανε και να περάσουμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 11 που θα ζητηθεί το πολύ μέχρι τις 5.30 γιατί στις 5.30 έχουμε κοινή συνεδρίαση με τις Επιτροπές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την ε, Επιθετιστική ασφάλεια στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας διατροφής για το 2015. Ελπίζω να δώσετε το παρόν στην κοινή αυτή συνεδρίαση των τριών επιτροπών. Γιατί δεν θα πρέπει να μείνουμε απόντες αυτή την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής ΔΕΒΕ θα πρέπει και εμείς να δώσουμε το παρόν ως μέλη της Επιτροπής ε, Γεωργίας. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας καλώ να περάσουμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 11, που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με θέμα τα δικαιώματα επιφυτικής ποικιλία των καλλιεργητών των φυτών και μια πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης φυτικών χαρακτηριστικών με δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Θα συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα των δικαιωμάτων των καλλιεργητών των φυτών, δικαιώματα φυτική ποικιλία. Ο συντονιστή για τα θέματα αυτά είναι ο κύριος Γιάνν Χόιτεμα από του μετά από την πρόσφατη απόφαση του Διευρυμένου Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Η απόφαση αυτή θα έχει σημαντικές συνέπειες για την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων και την ασφάλεια την επισητιστική. Οι συντονιστές πρότειναν να διεξαχθεί συζήτηση στην σημερινή συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Έχουμε εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται ακριβώς με το θέμα αυτό Θα δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Χέιτεμα για να μας παρουσιάσει αυτό το θέμα και να μας εκφέρει και τις απόψεις του γιατί ήταν δική του πρωτοβουλία και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ακολουθήσει συζήτηση γύρω σε ερωταπαντήσεων. Παρακαλώ κύριε Χαϊτεμα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα και θα μιλήσω Ολλανδικά. Θα ξεκινήσω καταρχήν ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους οι οποίοι με υποστήριξαν και θέλησαν μαζί μου να μπει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Στις 25 Μαρτίου το γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αναφέρθηκε μετά από την έφεση κατά της απόφασής του στο θέμα της δυνατότητας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για κάποια συγκεκριμένα φυτά, ποικιλίε φυτών. Το 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη είχε προετοιμάσει μια έκθεση με το θέμα αυτό και έφτασε σε κάποια συμπεράσματα όπως ζήτησε από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας να κρατήσει τις συμβατικές τεχνικές όσον αφορά τα δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λέγοντας ότι ε, πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματα των καλλιεργητών. Αυτή ήταν το 2012 η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά την απόφαση αυτή του Γραφείου Διπλωμάτων Ευαισθητεχνίας τίποτα απολύτως δεν έγινε. Τα δικαιώματα των καλλιεργητών, των παραγωγών θα πρέπει βεβαίως να βρίσκεται από τη μία λαμβάνοντας υπόψη την προστασία αυτών των δικαιωμάτων αλλά βεβαίως ε, την, ε, μη περιορίζοντας την ανάπτυξη. Είναι απαραίτητο αυτό γιατί πρόκειται για την ε, ασφάλεια των, ιδιών, των ειδών διατροφής και βάσει των πορισμάτων της ΦΑΟ έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά οι ποικιλίε και σήμερα βλέπουμε ότι 30 ποικιλίε είναι αυτές που καλύπτουν πάνω από το 95% της παραγωγής. Βλέπουμε λοιπόν ότι μειώνονται οι ποικιλίε και παραδείγματο χάρη μία ασθένεια, μία επιδημία θα είναι καθοριστική, μπορεί να αποτελέσει μάστιγα και να θέσει σε κίνδυνο την ε, ασφάλεια πολλών ποικιλιών, εκατοντάδων ποικιλιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα υπάρχουν 200 αιτήσει για διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φυτά, κυρίως για λαχανικά. Οι αιτήσει για άδειε ε, σαφώς και θα αυξηθούν. Αυτή είναι η τάση και γι' αυτό και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ να δράσει. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να πιέσω προς αυτή την κατεύθυνση. Κάνω μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα αυτά, ιδιαίτερα για τις συμβατικές ε, τεχνικές. Ζήτησα λοιπόν να μπει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και για να μην υπάρχει καμία απολύτως ε, παρερμηνία, σκοπός μου δεν είναι να ανοίξω το κουτί της Πανδώρας για την οδηγία σε θέματα που άπτονται της οδηγίας ε, για την βιοτεχνολογία. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θέλω να περιορίσω κάποιες νέες τεχνολογίες, αλλά είναι σημαντικό να εντοπίσουμε ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά κάποιων φυτών, κάποιων ποικιλιών που μπορεί να αποτελέσουν απελή για τις υπόλοιπες ποικιλίε. Και γι' αυτό και μιλάμε για εφεύρεση και όχι για ανακάλυψη. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ζανλίκ Γκάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε κύριε Χόιτεμα και ευχαριστώ και τους Ευρωβουλευτές και την Επιτροπή σας για την ευκαιρία που μας δίνετε και τη δυνατότητα να σχολιάσουμε αυτή την επικάλυψη μεταξύ διπλωμάτων ευρυστεχνίας και των δικαιωμάτων επιφυτικής ποικιλία. Ε, το διευρυμένο Προεδρείο του ε, Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρωπαϊκής το Μάρτιο ε, εξέδωσε μία απόφαση για τα φυτά που προκύπτουν από βιοτεχνολογικές διαδικασίες. Βέβαια πρόκειται για μία ανεξάρτητο οργανισμό το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία που εξέδωσε αυτή την απόφαση δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φυσικά υπάρχουν πολιτικέ συνέπειε τη απόφαση του γραφείου αυτού. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα του θέματο και παρακολουθούμε προσεκτικά και εκ του σύνεγγυ ε, την έκβαση αυτή τη απόφαση. Βέβαια και οι καλλιεργητέ ε, συγκεκριμένων χωρών μάλιστα μα ε, διαμήνυσαν τα προβλήματά τους και τις ανησυχίες τους και γνωρίζουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θυμάται κάλλιστα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2012 για το συγκεκριμένο θέμα και γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήσε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων Μία ομάδα εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από 15 εμπειρογνώμονες ε, με διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές καταγωγής. Δεν πρόκειται μόνο για ε, ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ε, είχαμε και εμπειρογνώμονες που δεν ήταν υπέρ της προστασίας από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Και εξετάζεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως αυτό που καλύπτει από την οδηγία. Ένα από τα θέματα που εξετάζει η ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων είναι αυτή η δυνατότητα κάλυψη με δίπλωμα ευρυστεχνία ε, φυτών που προκύπτουν από βιοτεχνολογικές διαδικασίες. Συνεχίζει η ομάδα εμπειρογνωμόνων το έργα τη ε, και περιμένουμε τα συμπεράσματά τους σε αρχές του επόμενου έτους επί Ολλανδικής Προεδρίας κατά πάσα πιθανότητα. Και φυσικά ε, θα δημοσιεύσουμε την γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας χάρη διαφάνειας και επίσης σας παραπέμπω και στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δείτε τη σύνθεση ακριβώς ε, της ομάδας των εμπειρογνωμόνων και να μελετήσετε και τα πρακτικά των συνεδριάσεών της αν σας ενδιαφέρουν. Οπότε θα εξετάσουμε φυσικά με προσοχή τις ε, συστάσεις των εμπειρογνωμόνων για να δούμε τι βήματα θα πραγματοποιήσουμε από εδώ και πέρα. Όπως είπατε σωστά, το ζήτημα είναι αρκετά επίγον και δεν περιμένουμε μόνο τη γνώμη και την απόφαση των εμπειρογνωμόνων. Εξετάζουμε και βραχυπρόθεσμες λύσεις, ώστε να ικανοποιήσουμε τουλάχιστον τους ενδιαφερομένους. Μία από τις ιδέες που έχουμε είναι να έχουμε από κοινού προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρυστεχνία και του Γραφείου για τα Δικαιώματα το Επιθετική Ποικιλία, ώστε να υπάρχει ένα συντονισμό κατά τη χορήγηση διπλωμάτων ευρυστεχνία. Γιατί αυτό το διευρυμένο ε, Προεδρείο για, την, για τις προσφυγές των διπλωμάτων ευρυστεχνίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια της καινοτομίας και της εφευρετικότητας ακριβώς επειδή το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Χέτεμα είναι θεμελιώδης, ένα τμήμα του ίσως ε, θα ε, επιληθεί με μια καλύτερη αξιολόγηση χάρη σε αυτή τη συνεργασία μεταξύ των δύο γραφείων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και σας ζητώ συγγνώμη κύριε Γκάλ που ξέχασα να αναφέρω το ονοματεπώνυμό σας πριν. Είστε από την Γενική Διεύθυνση Grow. Σας καλωσορίζουμε θερμά λοιπόν στη συνεδρίασή μας κύριε Γκάλ. Δίθεν το λόγο μερικοί ευρωβουλευτές. Πρώτη κυρία Ράνς Γκαρσία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντηση. Πάνω απ' όλα όμως ευχαριστώ τον κύριο Χέιτεμα που ανέλαβε την πρωτοβουλία να θέσει προς το θέμα αυτό. Θα ήθελα να είναι σαφή η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, γιατί αν ακριβώς είχαμε ένα... Ε, έχουμε, αν έχουμε ένα τομέα καινοτομία είναι ακριβώς αυτών των καλλιεργητών, των φυτών και των ε, σπόρων. και αυτό πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί από το 69 χάρη στην σύμβαση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τις φυτικές ποικιλίε, καταφέραμε να έχουμε την ανάπτυξη βιοτεχνολογίας και το έμας με μάση. Με την πρόσφατη όμως απόφαση του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας διακυβεύεται η εξέλιξη αυτή στο μέλλον. Η Οδηγία 44 του 98 δεν συνάδει με τις αρχές της Σύμβασης της ε, Ένωσης ε, Διπλωμάτων Επιστεχνίας για τις φυτικές ποικιλίε και των διαδοχικών τροπολογιών τη σύμβαση. Αν τώρα με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Επιστεχνίας θα έχουμε αυτά τα trades, ε, ακόμη και τα βιολογικά να μπορούν να καλύπτονται από διπλώματα ευρυστεχνίας, δηλαδή ακόμη και τότε που δεν υπήρχε η βιοτεχνολογία να υπάρχει δυνατότητα χορήγηση διπλωμάτων ευρυστεχνίας, τότε θα μπορεί να θα δοθεί δικαίωμα να καλύπτεται από δίπλωμα ευρυστεχνία σε οποιοδήποτε γονίδιο. Ακόμη και γονίδιο θα ζητάνε οι επιχειρήσεις να καλύπτονται από διπλώματα ευρυστεχνίας και, και να εμποδίζουν τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να το χρησιμοποιούν. Εμείς ε, με τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των γονιδίων δώσαμε μεγάλη ε, πολλές ευκαιρίες στη βιοτεχνολογία. Αλλά με την ε, τελευταία απόφαση δημιουργείται μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση. Είναι σαν να εμποδίζουμε την ιδιωτική, τη δημόσια πρωτοβουλία, την ε, δημόσια και την ιδιωτική έρευνα να προχωρήσουν. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Επιστεχνίας δεν θα πρέπει να δημιουργεί προσκόμματα και να παρεμποδίζει την ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Γιατί λέμε ναι στα διπλώματα ευρυστεχνίας, αλλά λέμε ναι και στην έρευνα. Και θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι δελαστική έρευνα και ελκυστική και για το δημόσιο τομέα και για τον ιδιωτικό. Δεν μπορεί το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρυστεχνίας να παρεμποδίζει αυτή την έρευνα. Προσοχή λοιπόν, γιατί θα κληθούμε να λάβουμε σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που είτε θα δώσουν ενάψματα στον ε, ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο να συνεχίσουν τις παιδί στην καινοτομία ή θα σκάψουμε μόνοι μας το λάκκο μας παρεμποδίζοντας αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Χόισλινγκ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ πολλές φορές δεν συμφωνούμε ιδεολογικά, αλλά νομίζω ότι εδώ και με άλλους συναδέλφους ξεκινήσαμε ένα κοινό ψήφισμα πριν από 4-5 χρόνια, το οποίο ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία εδώ και λέγαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίπλωμα τεχνίας επί ζώντων οργανισμών για τη ζωή. Και επικρίναμε τότε την προσπάθεια πολλών να καλύψουν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας οργανισμούς ε, που ήταν βεβαίως αποτελέσματα διαργασιών της βιοτεχνολογίας και νομίζω ότι και εδώ υπάρχει κάτι σε αυτήν την ε, σημερινή συζήτηση που θα πρέπει να μας οδηγήσει στο ίδιο συμπέρασμα. Άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως ε, καταλαβαίνω ότι το γραφείο διπλωμάτων ευαισθητεχνίας δεν είναι ένας αυτόνομος οργανισμός που λειτουργεί μόνος του οι αποφάσεις σαφώς και θα πρέπει εδώ να ισχύουν για όλους και να γίνονται πράξη κάτι που σήμερα νομίζω δεν μας διασφαλίζει η υπάρχουσα κατάσταση. Το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ουσιαστικά ζει από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αδειοδοτεί και που εγκρίνει. Είναι ο λόγος ύπαρξής του. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε λίγο το ερώτημα που αρχικά θέσαμε στην Επιτροπή. Είμαστε πολύ συγκεκριμένοι όσον αφορά το προηγούμενο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και επαναλαμβάνω ότι ο σημερινός μας η σημερινή μας κατεύθυνση σε αυτή τη συζήτηση δεν νομίζω ότι θα αποκλίνει πολύ από εκείνη που είχαμε πριν από 4-5 χρόνια. Και θα πρέπει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εμπειρογνώμονές της να αξιολογήσουν αυτά που συμβαίνουν. Θα πρέπει εδώ να προστατεύσουμε αυτήν την διαδικασία κάλυψης με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και όχι μόνο βεβαίως για τα φυτά. Πιστεύω ότι εδώ και άλλες ευρωπαϊκές και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές θα εμπλακούν και νομίζω ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε όλοι προς κοινά συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο Φρίδομ στον 19ο αιώνα έλεγε ότι η ευρεσιτεχνία είναι κλοπή, η κατοχή, συγγνώμη, η ιδιοκτησία είναι ε, κλοπή. Εγώ δεν θα φτάσω μέχρι εκεί. Παρ' όλα αυτά, ε, τον Μάριο του 2015, υπό την προεδρία του κυρίου Τωμά, με την απόφαση, το εφεσιδικείο της ε, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρωσιτεχνίας ε, απεφάνθη ότι ε, δεν είναι δυνατόν οι άγριες φύτρες να θεωρηθούν αντικείμενο ευρεσιτεχνίας και σύμφωνα με το άρθρο αλλά και με το άρθρο 54 ε, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Συνθήκη Λειτουργίας του Γραφείου Ευρεσιτεχνίας που λέει ότι οποιαδήποτε, ε, ε, οποιαδήποτε ζώσα μορφή είτε σε ζώα είτε σε φυτά εμπροκειμένο δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει να κατοχυρωθεί με ευρεσιτεχνία και εν πάση περιπτώσει δεν είναι δυνατόν αυτή να υπάρχει εσαΐ. Οπωσδήποτε εδώ θα πρέπει να ληφθεί κάποια κάποια ε, απόφαση συγκεκριμένη ε, γιατί εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο αίτημα ε, και περιμένουν ακόμα οι 200 περιπτώσεις όπως υπόθηκε προηγουμένως. Επομένως θα πρέπει η Κομισιόν να αποφανθεί. Εγώ μάλιστα είχα υποβάλει και ερώτημα την 23η Ιουνίου στην Κομισιόν, δεν είχε απαντηθεί ακόμα, μεσολάβησαν βέβαια διακοπές κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε θα πρέπει ε, να, ε, να, να ξαναδούμε λίγο την 4498 ε, έτσι ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε ιδιοποίηση του δημοσίου τομέα που εκεί όντως ισούται με κλοπή. Κύριε Πρόεδρε, όταν ε, ο Μάρτιν Χάουσλινγκ και εγώ συμφωνούμε σε κάτι, τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να υποκληθεί η Κομισιόν. Δεν συμβαίνει αυτό κάθε μέρα. Ε, όντως εδώ δημιουργείται προηγούμενο γιατί ε, ε, ε λέμε ότι μπορεί να κατοχυρωθεί ένα χαρακτηριστικό αλλά όχι όμως η ποικιλία από την οποία προκύπτει το χαρακτηριστικό αυτό. Τρία είναι τα σημεία τα οποία ε, ε, δημιουργούν πρόβλημα. Είναι ένα ηθικό ζήτημα, ζήτημα δεοντολογίας, ε, διότι αναφέρεται σαφώς ότι δεν είναι δυνατόν ζών οργανισμός να αποτελέσει αντικείμενο κατοχήρωσης και εμπορίας. Δεύτερον, δεν γίνονται σαφή πλέον με τον τρόπο αυτό τα όρια μεταξύ εφεύρεσης και ανακάλυψης ε, και στην ουσία εδώ δυσκολευόμαστε χωρίς λόγο. Τρίτον, ε, η Κομισιόν λέει ότι υποσκάπτεται με τον τρόπο αυτό η ελεύθερη δυνατότητα ανάπτυξης νέων χαρακτηριστικών ε, νέας επομένως στρατηγικής που μπορεί να οδηγήσει και σε εμπορική στρατηγική. Δεν το θέλουμε λοιπόν αυτό. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα από το παρελθόν όταν η Γεωργία ε, στην ουσία χρησιμοποιούσε ε, τα απλά χαρακτηριστικά. Ε, νομίζω ότι χρησιμοποιήσαμε τις ε, σκληρές στήλες στους πασάλους για να κρατάμε ε, τα φυτά τα οποία διαφορετικά με τον αέρα θα έπεφταν. Αυτό είναι, θα χάναμε σε ποιότητα, θα χάναμε σε ποσότητα ε, και βρήκαμε λοιπόν το, το, το, σκληρό μισχοσιτάρι. Ε, νομίζω ότι αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο κατοχύρωσης γιατί διαφορετικά θα είχαμε πρόβλημα σε αναφορά τη γενοτομία και τη χρήση της καινοτομία. όλοι θα χρησιμοποιούσαν ακριβώς τα, τις ίδιες ε, ε, φυλές ε, και θα είχαμε πρόβλημα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, όταν κάποιος βρίσκει κάτι ε, ε, ή κάποιος ο οποίος ε, ανακαλύπτει ας πούμε ή χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο κάτι το οποίο υπάρχει στη φύση θα πρέπει να, να μπορεί να το πατεντάρει και να το χρησιμοποιήσει μετά να βγάλει χρήματα από την πατέντα αυτή. νομίζω ότι θα πρέπει η Κομισιόν να μην κάνει τίποτα που να μπορεί να μπλοκάρει οποιαδήποτε καινοτομία. Dziękuję. Pan poseł Dorfman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έφερε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως συμφωνώ με τους περισσότερους ε, όπως πήραν το λόγο μέχρι τώρα. Να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην μπερδέψουμε την προστασία κάποιων ειδών, κάποιων ποικιλιών, αλλά την, με την δυνατότητα κάλυψης τους από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Και εδώ θα πρέπει να ισχύσει το υπάρχον δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να διευρύνουμε την προστασία των δικαιωμάτων για τις ε, αν θέλετε, συναλλαγές ε, και αυτό που είναι σημαντικό όσον αφορά την κάλυψη από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι η δυνατότητα καλλιέργειας. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πρέπει, συγγνώμη, ο καθένας θα πρέπει να μπορεί να καλλιεργήσει, να επιλέξει ε, μία ποικιλία και αν υπάρξουν περιορισμοί αν δηλαδή δεχτούμε την δυνατότητα κάλυψης από διπλώματα ευρεσταχνίας κάποιων ποικιλιών, είναι σαν ουσιαστικά να αφήνουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, μόνο τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, να ε, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά. Οι μικροί καλλιεργητές θα εξαφανιστούν. Σήμερα, όπως ξέρετε, υπάρχουν πολύ λίγα, πολύ λίγοι σπόροι, πολύ λίγες ποικιλίε που είναι προϊόντα βεβαίως πολύ συγκεκριμένων τεχνικών που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ξέρουμε ποιος τα διαθέτει, ποιος τα καλλιεργεί και ποιος τα πολύ τελικά. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε τους καλλιεργητές, τους παραγωγούς, κυρίως τους πιο αδύναμους και καταλαβαίνει πολύ καλά η Επιτροπή ότι η αγορά θα αλλάξει άρδιν αν κάτι τέτοιο συμβεί και αν υποχωρήσουμε. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση, πολιτική πίεση, για να μην γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε Πετήρ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, γιατί ήρθαν σε επαφή μαζί μου πολλοί καλλιεργητές και δημιουργοί νέων ποικιλιών και εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών που είναι κατά τη απόφαση αυτή, ε, γιατί φοβούνται τι συνέπειε που θα έχει μια τέτοια απόφαση του Γραφείου Προσφυγών ε, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία. Έχει ένα μικρό πρόβλημα με την κρατική διερμηνία. Συνεχίζουμε τώρα. Όπως είπα, ήρθαν σε επαφή μαζί μου πολλοί καλλιεργητέ ε, και δημιουργοί νέων ποικιλιών, αλλά και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, που είναι ενάντια στην απόφαση αυτή, γιατί φοβούνται τις ε, συνέπειες, τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει για τον κλάδο, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες με τους οποίους συμφωνώ. Επίσης, μια τέτοια απόφαση του Γραφείου Προσφυγών ε, θα καταστρέψει το οικονομικό δυναμικό των ε, δημιουργών νέων ποικιλιών και των καλλιεργητών. Γιατί θα αυξήσει το κόστος και είναι και απρόβλεπτο το πόσο τελικά θα αυξήσει το κόστος αυτών των διπλωμάτων τεχνίας. Επίσης φοβούνται και τη μελλοντική συγκέντρωση που θα παρουσιαστεί στην αγορά σπόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιου είδους αποφάσεις όλο και περισσότερες πολυεθνικές ε, θα προσπαθούν να καρποθούν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς των σπόρων. Είναι λοιπόν κατά της, ε, για ηθικούς λόγους ε, της χορήγης διπλωμάτων ευρυστεχνία σε ζωντανούς οργανισμούς. Δεν μπορούμε να καλύπτουμε με δίπλωμα ευρεσιτεχνία στη ζωή τα ζωντανά πλάσματα. Και σίγουρα θα πρέπει να γίνουμε έρμεο των πολυεθνικών. Θα πρέπει να σταματήσουν οι πολυεθνικές να παίζουν τον Θεό πολλές φορές. Συμφωνώ λοιπόν με την πρωτοβουλία του συναδέλφου Χόιτεμα και το συγχαίρω για την πρωτοβουλία του, γιατί μετά από την απόφαση αυτή ε, χιλιάδες ε, αιτήσει για διπλώματα βριστεχνίας που μέχρι στιγμής ε, είχαν απορριφθεί γιατί ήταν απαγορευμένες, ε, ανοίγεται πιο ο δρόμος να εγκριθούν. Θα πρέπει λοιπόν να απαγορεύσουμε τέτοιου είδους αποφάσεις, δηλαδή δυνατότητες να καλύπτονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, ζωντανοί οργανισμοί, είτε φυτών είτε ζώων και ε, παραπέμπω στο άρθρο 4 της οδηγίας 48 ε, του 99 και περιμένουμε μια ανάληψη δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Μπέλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι ανησυχώ γιατί η υπηρεσία, ε, το Γραφείο Ευρεσιτεχνίας μάλλον, επιβεβαίωσε αυτήν την ε, απόφαση. Είναι κάτι το οποίο ε, δεν είχε προβλεφθεί από την νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να καλυφθεί το κενό αυτό. Το 2012 το Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει μια ε, ε, έκθεση ε, πολύ ισχυρή κατά των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Θα πρέπει πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει για μία ακόμα φορά να στραφούμε προς την Επιτροπή κατά την έννοια αυτή που μόλις ανέφερα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σένερα. Δεν μας έχουν μείνει και πολλά επιχειρήματα πια. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω την κάθετη αντίθεσή μου σε αυτή την απόφαση να δίνονται διπλώματα ευρυστεχνία για φυτικές ποικιλίε, για φυτά. Θα ήθελα να μα εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τι γίνεται με αυτό το πιλωτικό σχέδιο που ανήγγειλε μεταξύ του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρυστεχνία και του ε, Γραφείου Δικαιωμάτων ε, Φυτικών Ποικιλιών. Τι πιλωτικό πρόγραμμα ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν κατάλαβα καλά ότι υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Ακούσαμε όλους τους ευρωβουλευτές που είχαν ζητήσει το λόγο, οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζων Γκάλ, για να απαντήσει. Παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you to all the of the European Parliament who uh, just... Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ και όλους όσους έφρασαν την άποψή τους. Καταρχήν να σας θυμίσω ότι από το 2012 δεν νομίζω ότι απλώς περίμενε άπρακτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας υπενθυμίζω ότι τότε υπήρξαν κάποια εκκρεμή θέματα ενώπιον του, της υπηρεσίας προσφυγών και το υπόθεση μπρόκολι 1 και ντομάτα 1 για τα οποία αναφερθήκατε ουσιαστικά απέκλεισαν τη δυνατότητα του Γραφείου Διπλωμάτων Ευαισθητεχνίας από την ιαδήποτε κάλυψη με διπλώματα ευαισθητεχνίας. Δηλαδή, ιδιαίτερα προϊόντα τα οποία προέρχονται από βιοτεχνολογικές διαδικασίες και διαργασίες. Μέχρι το Μάρτιο που ελήφθη η απόφαση, αυτή ήταν η κατάσταση. Από τότε μέχρι σήμερα βέβαια δεν έχει περάσει πολύς ε, χρόνος. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων εργάζεται σκληρά, επεξεργάζεται τα διάφορα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και σήμερα μας ζητάτε τροποποίηση και αποσαφήνιση. Η απόφαση σίγουρα θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να μπορέσει να αποσαφηνίσει και δεν είναι εύκολο σήμερα να αλλάξει αυτή η νομοθεσία καθότι πρόκειται για νομοθεσία που διέπει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρυστεχνίας. Οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνονται με τρόπο συλλογικό. Εξετάζουμε λοιπόν βραχυπρόθεσμη απόφαση και αναφέρθηκα και στο πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο ενδεχομένω θα έχει σαν σκοπό να τεθούν προτεραιότητες, έτσι ώστε να μην δοθούν σε κάθε περίπτωση τέτοια ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εκτός εάν πρόκειται για καινοτόμα προϊόντα και βεβαίως σκοπός μας είναι στην πράξη να βελτιώσουμε την κατάσταση και να αποφύγουμε κάθε είδους δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε αυτό το τομέα. Γιατί όντως υπάρχει πίεση για αύξηση του αριθμού. Πρόκειται λοιπόν καταρχήν για ένα θέμα αρχής. Αν ναι ή όχι, μπορεί να δοθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα προϊόν το οποίο προέρχεται από μια βιολογική, βιοτεχνολογική διαδικασία. Και η απόφαση αυτή θα ληφθεί, πιστεύω, ε, μόλις ολοκληρώσει η αρμόδια επιτροπή της εργασίας της. Θα δώσω τώρα τον λόγο στη συνάδελφο από την DG Sante. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας καθησυχάσω. Παρακολουθούμε στενά αυτό το θέμα, καθώς και τις αποφάσεις ε, της υπηρεσίας προσφυγών του Γραφείου Διπλωμάτων Τεχνίας όσον αφορά τα θέματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των ε, παραγωγών, των καλλιεργητών και φυσικά την προστασία των ποικιλιών. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, καθότι τα προϊόντα αυτά βρίσκονται στην καρδιά της διατροφικής αλυσίδας. Θέλουμε μια πιο πράσινη οικονομία και σε κάθε περίπτωση επιθυμούμε να προστατεύσουμε τον τομέα αυτό οργανώσαμε και ένα σεμινάριο με εμπειρογνωμόνες. Η συζήτηση που έγινε στα πλαίσια αυτά ήταν πολύ επικοδομητική. Ακούστηκαν πολλές απόψεις για την δυνατότητα κάλυψης με διπλώματα βρεστεχνίας, για ποιες ποικιλίε. Βεβαίως υπάρχει και βραχυπρόθεσμα ανάγκη για απόφαση, αλλά χρειάζεται ακόμα εργασία, συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Αυτό έχει ξεκινήσει και από ό,τι φαίνεται το πιο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί ένα κείμενο Prior Act να υπάρχει πρόσβαση τα δεδομένα και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα απαιτηθούν αυστηρότερα πρότυπα και δεδομένα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που αφορούν τις ποικιλίε των φυτών. Σας ευχαριστώ. Θέλει πως ο κύριος Χαϊτεμα να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους γιατί φάνηκε ευρία συνένεση και σύμπνοια μεταξύ μας. Όλοι θεωρούμε πολύ σημαντικό το θέμα και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους και καλό θα ήταν ίσως να εκπονήσουμε και να ψήφισουμε. γιατί είχαμε ήδη ψηφισμό στο παρελθόν, καταθέσαμε και προφορική ερώτηση ε, και να παραλάβουμε μια προφορική ερώτηση με ψήφισμα για να ασκήσουμε πολιτική πίεση, γιατί το θέμα όντω είναι πολύ σημαντικό. Okay możemy Καλώς. Οπότε ολοκληρώνουμε αυτό το θέμα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Χαίτεμα για την πρωτοβουλία που ανέλαβε να θέσει προς συζήτηση αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Πολύ σημαντικές ε, συζητήσεις είχαμε για την κρίση, για την μεταρρύθμιση ε, της ΚΑΠ, αλλά λίγο ασχολούμαστε με τέτοια θέματα που θα αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον. Γιατί η δημιουργία νέων ποικιλιών είναι πολύ σημαντικό θέμα και φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση δημιουργίας μονοπωλίων και συγκέντρωσης. Κάτι που απειλεί και τους παραγωγούς, ε, τους γεωργούς, αλλά απειλεί και τους ίδιους τους καταναλωτές. Δημιουργεί κίνδυνο και για αυτούς. Και φαίνεται ότι επικρατούν τα εμπορικά επιχειρήματα στο θέμα της δημιουργίας νέων ε, ποικιλιών, κάτι που επηρεάζει αρνητικά ολόκληρο τον κλάδο. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σταθεί στο πλευρό των γεωργών και να προασπίσει τα δικά τους συμφέροντα. Γιατί οι γεωργοί δεν έχουν την ισχύ που έχουν στην αγορά οι πολυεθνικές, οπότε είναι ανήμποροι απέναντι τους. Γι' θα πρέπει να τονίσουμε την υποστήριξή μας προς την καινοτομία, προς την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και κυρίως την υποστήριξή μας προς τους μικρούς παραγωγούς και καλλιεργητές που δεν θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα. Εξίσου σημαντικό με τα άλλα πολύ σημαντικά που συζητήσαμε και χαίρομαι γιατί φάνηκε ευρεία συνένεση μεταξύ μας για το θέμα αυτό. Οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα ήταν να, να το λάβει σοβαρά υπόψη. Εμείς σίγουρα θα επανέλθουμε γιατί οι αποφάσεις μας θα επηρεάσουν την καινοτομία και κάποιες αλλαγές που θα χρειαστούν για να εξασφαλίσουμε την επισητιστική ασφάλεια, την ασφάλεια των τροφίμων. Σας ευχαριστώ θερμά. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Την έγκριση των συστάσεων που εξέδωσαν οι συντονιστές. Ο κύριος Νίκολσον. Ναι. Στις τελευταίες σελίδες να βρω λίγο τα χαρτιά μου, ή τα χασά, λέει ο κύριος Νίκολσον. 7.2. Uh, το 7.2. Στο 7.2 λοιπόν, στην προτελευταία γραμμή, ε, να βγουν, το, ε, να βγουν ε, οι λέξεις impossible to Terry. Okay, bardzo proszę autora. Παρακαλώ την γραμματεία που συνέταξε για το κείμενο. Ναι, ωραία, θα κάνουμε αυτή τη διόρθωση από τη στιγμή που δεν φαίνεται κανείς να αντιτίθεται σε αυτό που μόλις είπα. Ωραία, Έγκριμε λοιπόν τη στάση των συντονιστών. Και μια παράκληση θερμή. Ελάτε στην ώρα σας, δηλαδή 5.30 και λίγο νωρίτερα γίνεται, στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών ΔΕΒΕ, ΕΜΒΙ και Άγκρη στην, ε, στον τρίτο όροφο, στην αίθουσα C50, στο κτίριο Polaris Park. Ήδη στις 5.30 να είμαστε όλοι εκεί παρακαλώ. Θα, δώσουν, θα λάβουν το λόγο οι συντονιστές για ένα λεπτό, αλλά θα έχουν την ευκαιρία και οι ευρωβουλευτές να λάβουν το λόγο σε αυτή την κοινή συνεδρία των τριών επιτροπών. Αυτά λύεται η συνεδρίαση. Έχουμε μάλιστα και διάλειμμα μία ώρα σχεδόν μέχρι την έναρξη της κοινή μας συνεδρίασης. Παρακαλώ, ελάτε όλοι στην 350 στο Polaris Park στις 5.30. Γεια σας.